Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι. Για ακούστε με σας παρακαλώ. Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής. Μπορείτε να μην κοιτάξετε. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας που Καθυστερούμε με την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης. Τελειώσαμε αργά την πρωινή συνεδρίαση, λόγω της ε, συζήτησης βέβαια με τους προσκεκλημένους μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν τώρα. Έχουμε τώρα τους προσκεκλημένους μας πάλι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και το αντικείμενο της ακροάσεως είναι αξιολόγηση της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την εμπορική πολιτική. Βέβαια, η ίδια η Επιτροπή θα συνεχίσει να δρά και να λειτουργεί μέχρι τον Οκτώβριο, νομίζω έτσι, με περιορισμένες κάπως ε, δραστηριότητες. Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει συντελεστεί μέσα στην πενταετία αυτή και σχεδόν ολόκληρη υπό τη συνθήκη υπό την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποίησε βέβαια σημαντικά την θεσμική ισορροπία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου των Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήρθε η ώρα λοιπόν, όπως έλεγα, να προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση για το τι έχει επιτευχθεί ποια πράγματα δεν πέτυχαν και βέβαια και την άποψη των ενδιαφερομένων, των stakeholder. Γιατί ο τομέας του εξωτερικού εμπορίου είναι σημαντικός. Ευχαριστώ και πάλι και ο Πασκάλ Σερνάης από το European Services Forum είναι επίσης ε, παρόν, ο κ. Χέντριξ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, ο κ. Νικολάη Σουκούπ της, του Αυστριακού μάλλον Ομοσπονδίας Εργασίας και η κυρία Κάριν Ούλμερ από την Απροντεύ. Έχει σχέση βέβαια με τις οργανώσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό αξιολογεί τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Εμείς βάλαμε επίτηδες υπέρ και κατά, αλλά νομίζω ότι στην αξιολόγησή σας εσείς δεν έχετε καθόλου και κατά. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Λέει ο κύριος Ντεμαρτή. Ας είμαστε μετριόφρονες, ακόμη και Βεβαίω όταν προσπαθούμε να επιτύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε καθηγητά και αξιότιμοι ευρωβουλευτές που διοργανώσατε την ακρόαση και όπου όντως είναι έγκαιροι τώρα στην αρχή έχω να τονίσω δύο πράγματα για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αντίθεση με τα παλαιότερα χρόνια, όχι μόνο ανοίξαμε νέες διαπραγματεύσεις, αλλά καταφέραμε και οδηγήσαμε και σε αίσιο πέρας πολλές διαπραγματεύσεις και αρχίσαμε την εφαρμογή νέων συμφωνιών. Διότι ωραία είναι να ανοίγει κανείς διαπραγματεύσεις, αλλά ο στόχος είναι και να τις ολοκληρώσει κανείς και να τις εφαρμόσει εποφελία των Ευρωπαίων πολιτών, να υπάρξει δηλαδή ανάπτυξη και απασχόληση. Δεύτερο, το μέγεθος της εμπορικής μας ατζέντα δεν έχει προηγούμενο και μάλιστα με τόσες διαπραγματεύσεις τις οποίες χειριζόμαστε ταυτόχρονα με σημαντικούς εταίρους με βιομηχανικές χώρες όπως τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις Ενωμένες Πολιτείες και μάλιστα και περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν η εμπορική πολιτική αποτελεί σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να οδηγεί στην οικονομική ανάκαμψη. Ως αποτέλεσμα η εμπορική πολιτική προσελκύει, προσελκύει βεβαίως τώρα πολύ περισσότερο την προσοχή. Τρία θέματα τώρα. Πρώτο, τι έχει επιτύχει το εμπόριο. Δεύτερο, την αύξουσα σημασία της αναπτύξεως στο έργο μας. Και τρίτο, τις αλλαγές που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρώτο, για τα όσα επιτύχαμε. Το ιστορικό είναι θετικό και αναφέρομαι πρώτα στην Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέας με Κολομβία, Περού και Κεντρική Αμερική. Με την Κορέα η συμφωνία είναι θετική για την Ένωση διότι οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών μας στην αγορά της Κορέας. Χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, σας λέω ότι οι εξαγωγές μάσης προς την Κορέα αυξήθηκαν κατά 24% ή 7 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας συγκριτικά με το πρώτο χρόνο που ήταν 2011 και επίσης η εξαγωγή αυτοκινήτων από την Ένωση στην Κορέα, το πιο δύσκολο μέρος της συμφωνίας αυτής, αυξήθηκε κατά 40% σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο. Επίσης, οδηγήσαμε σε τελική φάση της ε, διαπραγματεύσεις με τη Σιγκαπούρη καθώς και με τον Καναδά. Επίσης βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για μείζονες συμφωνίες με τις Ενωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία καθώς και με την Κίνα. Αυτά είναι σημαντική διαφορά ανάμεσα στα όσα συνέβαιναν πριν από τέσσερα χρόνια και στοχεύουμε και σε άλλες συμφωνίες με άλλες χώρες της ε, Ασίας αλλά και με την νότια πλευρά της Μεσογείου. Έχουμε μετακινήσει τώρα την στόχευσή μας από τις πολυμερείς συμφωνίες σε διμερείς συμφωνίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τις ευεργετικές επιδράσεις των πολυμερών συμφωνιών και του ΠΟΕ μας επιβλήθη από τις γνωστές συνθήκες η αλλαγή στόχευσης. Βεβαίως εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τις πολυμερείς συμφωνίες, το ίδιο όπως και εσείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ολοκλήρωση του γύρου του Μπαλί. Για πρώτη φορά λοιπόν τέτοια πολυμερή συμφωνία μετά από την ε, ίδρυση του, οργανισμού, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δηλαδή και ορισμένοι από εσά ήσασταν παρόντες στον Παλί. και με λήψη υπόψη ιδίω των συμφερόντων των αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης υπάρχουν πολυμερείς ε, πρωτοβουλίες για τον τομέα των υπηρεσιών καθώς και για τα πράσινα αγαθά με στόχο να γίνουν οι συμφωνίες αυτές πολυμερείς μακροπρόθεσμα. Ο στόχος παραδοσιακά των εμπορικών διαπραγματεύσεων είναι να ανοίξουν νέες αγορές για τις επιχειρήσεις και βεβαίως εξακολουθεί να ισχύει. 90% της μελλοντική ανάπτυξης θα σημειώνεται εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας βέβαια τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν να αναπτύξουμε το σύστημα του εμπορίου και στην ανακοίνωση του 2012 για το εμπόριο ανάπτυξη και αύξηση ήταν αυτός ο στόχος. Τώρα, παράδειγμα, έχουμε μεταρρυθμίσει το γενικό σύστημα προτιμήσεων. Στοχεύει τώρα σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Συνεχίσαμε τις ε, συμφωνίες μας με τις χώρες της Αφρικής, ιδίως της Δυτικής Αφρικής, με μια πολύ σημαντική συμφωνία στον Τακάρ την προηγούμενη εβδομάδα, με συμμετοχή του αρμόδιου επιτρόπου και βεβαίως και του Προέδρου Μακισάλ Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της παραμένουν και ο μεγαλύτερος δωρητής, δωρητής συγγνώμη, με 9,4 δισεκατομμύρια στο σύστημα Aid for Trade. Επαναλαμβάνουμε δε την δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνοντας σχετικά κεφάλαια στις συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε. Τέταρτο, μετά από την τραγωδία του Μπαγκλαντές, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και τις Ηνωμένε Πολιτείες κατέληξαν στη συμφωνία για το Παγκλαντές για την τήρηση των προδιαγραφών εργασίας και για την ανάληψη των ευθυνών της υφαντολογικής βιομηχανίας. Τέλος, σημαντικό επίτευγμα των τελευταίων τεσσάρων ετών ήταν και η προσπάθειά μας για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Προτείναμε να ολοκληρωθούν τα δύο πακέτα όμνιμπους για τις εκτελεστικές και κατεξουσιοδότηση πράξη πράξεις μεν, αλλά λιγότερο ίσως περιεκτικές από ορισμένες άλλες πολιτικές. Δεύτερο, αρχίσαμε να στείλουμε στα πόδια της μια νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επενδύσεις. Γνωρίζω ότι η άποψή σας για ορισμένα, ορισμένες από τις ευχές του θέματος είναι λιγότερο θετικές, αλλά τώρα προχωρούμε με τον σχετικό κανονισμό Κάναμε μια πρόταση για την οικονομική ευθύνη για τις σχέσεις επενδυτών με τα κράτη και δεν θα σταματήσουμε. Χρειαζόμαστε νέα, πιο ισορροπημένη προσέγγιση για την προστασία των επενδύσεων. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις επενδύσεων με την Κίνα και πρόκειται να πράξουμε το ίδιο και με την Μιανμάρ. Και όλες μας οι νέες συμφωνίες έχουν και ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Είναι αλήθεια βέβαια ότι η θέσπιση των πολιτικών αυτών δεν ήταν και εύκολη και ορισμένες χώρες μέλη εξακολουθούν να έχουν προβλήματα με το γεγονός ότι οι επενδύσεις μπαίνουν σε άλλη αρμοδιότητα. Ευτυχώς έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Και έρχομαι στο τελευταίο μου σχόλιο για την σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου, που κατά τη γνώμη μου υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής. Ίσως να μην συμφωνούσαμε πάντοτε, αλλά έχουμε πολλούς κοινού στόχους για την πολιτική εμπορίου. Και συχνά έχουμε συνεργαστεί με αμοιβαίο σεβασμό των θεσμικών μας ρόλων. Η δική σας συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων για την εμπορική πολιτική έχει αυξηθεί, επομένως και η διαφάνεια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στη θαυμάσια αυτή συνεργασία και στην επόμενη θητεία. Όσοι εξ ημών επανεκλεγείτε ευρωβουλευτές και θα επανέλθετε ενδεχομένω στην Επιτροπή Ίντα, μπορώ να σα υποσχεθώ ότι θα έχετε πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια για να υιοθετηθούν τα τελικά αποτελέσματα των προσπαθειών που έχουμε αναλάβει τα τελευταία χρόνια. Ως τελικό συμπέρασμα θα έλεγα ότι βεβαίως δεν επαναπαυόμαστε, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία στην ατζέντα, Πάντοτε βεβαίως μπορούμε να επιτύχουμε και κάτι παραπάνω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να υλοποιήσουμε όλα τα στοιχεία της ατζέντα που είναι ανοιχτή αλλά και πάρα πολύ μεγάλη, να τα ολοκληρώσουμε έγκαιρα, εποφελία των Ευρωπαίων πολιτών και πάλι για να υπάρξει ανάπτυξη και απασχόληση, διότι αυτά είναι που έχουν σημασία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια αυτή η δική μας επιτροπή θα είναι περιζήτητη. Επόμενος ομιλητής είναι ο Πασκάλ Κερνάης που είναι διευθυντής του, φόρουμ, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Υπηρεσίες. Καλά νέα Πασκάλ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Έχεις το λόγο. Ποια είναι η γνώμη σου για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο εδώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ συμμερίζομαι πολλές από τις απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Δημαρτή, γιατί πιστεύω πως η τούτη Επιτροπή κατάφερε να πετύχει εντυπωσιακά και συγκεκριμένα αποτελέσματα τα περισσότερα από αυτά τα ανέφερε ο κύριος Δεμαρτή, αλλά είναι σημαντικό να τα δούμε και σε σχέση με το τι έγινε σε προηγούμενες ε, ε, θητείες. Συνήφθησαν αλλά και εφαρμόστηκαν ε, πολλές συμφωνίες. Ο οργανισμός μας ε, δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσουμε κενά στον ΠΟΕ και έχουμε, είχαμε κολλήσει στο DDA εδώ και πολλά χρόνια και τώρα επιτέλους έχουμε κάποια αποτελέσματα. Δεν θα διαβάσω όλο τον κατάλογο γιατί δεν έχουμε το χρόνο, αλλά είναι ένας μακρύς κατάλογος πολύ εντυπωσιακών αποτελεσμάτων και πρέπει αυτό νομίζω να τονιστεί. Έχουμε ήδη, όπως είπαμε, την συμφωνία για το εμπόριο στις υπηρεσίες που είναι πολυμερείς διαπραγματεύσεις στη Γενέβη. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει 6 γύρους και 20 χώρες συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις αυτές. Ο επόμενος γύρος θα γίνει του χρόνου η ε, διευκόλυνση, η συμφωνία διευκόλυνση εμπορίου στον Παλί είναι κάτι πολύ θετικό επίσης. Θεωρείται πολύ συχνά ένα καλό θέμα γιατί πρόκειται για εταιρείε που περνούν τα σύνορα με τις οι υπηρεσίες τους ε, ε, είναι διάφοροι φορείς, κάτι πολύ ενδιαφέρον και είμαστε ε, ευχαριστημένοι που ανακοινώθηκε μια νέα συμφωνία για πράσινα αγαθά και ελπίζουμε πως όχι μόνο θα έχουμε τις τελωνιακές γραμμές για αυτά τα αγαθά αλλά και για τις υπηρεσίες και αν δεν συμβεί αυτό σε αυτήν την ομάδα θα μπορούσε να εξεταστεί τουλάχιστον σοβαρά στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ΤΙΣΑ. Τι μας προσέφερε λοιπόν αυτό, περισσότερη πρόσβαση στις αγορές, ε, έχουμε πιο συγκεκριμένη νέα πρόσβαση στην αγορά για τις ευρωπαϊκές εταιρείε υπηρεσιών στους ε, χρηματοπιστωτικό τομέα, στο νομικό τομέα, σε άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες, στις τηλεπικοινωνίες, στις ε, ναυτιλιακά Περιβαλλοντικέ υπηρεσίες και όλα αυτά τα έχουμε διαπραγματευτεί και έχουμε κερδίσει την πρόσβαση. Είναι αλήθεια πως είναι πιο περίπλοκο το να δούμε αποτελέσματα στο εμπόριο υπηρεσιών γιατί δεν έχουμε ισοζύγιο πληρωμών στο σύνορο οπότε είναι πιο περίπλοκο αλλά η αύξηση του εμπορίου σε υπηρεσίες στη διάρκεια των ετών είναι σαφή απόδειξη πω αυτέ οι νέε αγορέ έχουν ανοίξει για τις επιχειρήσεις μας. Επίσης έχουμε νέα πρόσβαση στις αγορές για τις δημόσιες προμήθειες, δημόσιες συμβάσεις όπου συχνά θεωρείται ένα θέμα αγαθών αλλά είναι και θέμα υπηρεσιών γιατί σε κάποιες χώρες έχουμε διαπραγματευτεί με την Ένωση για τοπικές ε, ή περιφερειακές ε, δημόσιες υπηρεσίες για δημόσια νοσοκομεία ή σχολεία όπου μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε στις, ε, στους διαχωρισμούς. Κινητικότητα είναι κάτι ακόμα για την ΓΚΑΤΣ επιτρέπεται δηλαδή οι εταιρείε να φέρουν κόσμο στις ε, θηγατρικές τους σε άλλες χώρες αλλά και τούμπαλιν γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε πως χρειάζεται να έχουμε εμπειρογνώμονες στις εταιρείε μας όταν αυτή είναι απαραίτητη. Επίσης αναφέρθηκε η προστασία των επενδύσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο, δεν έχουμε το τελικό κείμενο Τη ΣΥΤΑ, ε, πρέπει να ελεγχθεί και είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να έχουμε ισχυρή προστασία, θα επανέλθουμε αργότερα. Περισσότερη διαφάνεια τώρα για τους κανονισμούς. Αυτό προσπαθούν να το έχουν όλες οι εταιρείες και σε όλες τις ε, συμφωνίες για ελεύθερες συναλλαγές είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις εταιρείες. Νέα έμφαση στην πολυμερή συνεργασία. Πιστεύουμε πως αυτός είναι ο δρόμος, κυρίως με το TDIP. θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Ε, ας πούμε στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι ένας νέος τρόπος να εξετάζουμε την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων, δεξιοτήτων, αδειοδοτήσεων για τις ε, επιχειρήσεις, αντί να χρειάζεται δηλαδή οι εταιρείε μας να στραφούν σε δύο διαφορετικές αρχές, Εάν μπορούν να συνεργαστούν οι αρχές στην εποπτεία ή στην εχορήγηση κάποιες άδειε, για παράδειγμα, θα μπορούσαν όλα να πάνε πιο γρήγορα και ελπίζουμε πως αυτό θα συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Αυτά ήταν τα θετικά στοιχεία. Τώρα Μπαίνουν βέβαια ακόμα να γίνουν πολλά. Καταρχήν για μας είναι η ε, διαπραγματεύσεις ΤΙΣΑ, δηλαδή εμπόριο στις υπηρεσίες, γιατί εκεί έχουμε κολλήσει μέσω ε, των διαπραγματεύσεων για την ΚΑΤΣ, για την DTA και στην ουσία οι υπηρεσίε κρατώνται όμοιροι της γεωργίας και γι' αυτό και προσπαθούμε να πιέσουμε για τις ε, διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες στη Γενέβη και ανέκαθεν λέγαμε ότι θέλαμε να συμμετέχουν περισσότερες ομάδες, μεγαλύτερες μάλλον ομάδες, γιατί μέχρι εμείς Έχουμε φιλοδοξίες με τις ομάδες που υπάρχουν και θα μπορούσαμε να ξανασχεδιάσουμε κάποιες συγκεκριμένες ε, αρχές για συγκεκριμένους τομείς, αλλά θέλουμε και νέες χώρες. Η Κίνα χτύπησε την πόρτα για να μπει στην ομάδα των διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς οι φίλοι μας, ε, οι Αμερικανοί, δεν είναι πολύ πρόθυμοι γιατί δεν είναι βέβαιοι για το τι ακριβώς θα κάνει η Κίνα, αν θα συμμετέχει πραγματικά δηλαδή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι αφήστε τους να μπουν και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Δεν ανάγκη να ληφθεί απόφαση εκ των προτέρων, να τους αφήσουμε να διαπραγματευτούν για να δούμε αν θα είναι έτοιμοι να προσφέρουν κάτι συγκεκριμένο. Γιατί διαφορετικά εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μας χωρίς την Κίνα. Αλλά τουλάχιστον να είναι στις διαπραγματεύσεις, γιατί η Κίνα τώρα ε, ε, η Κίνα ε, εμποδίζει και άλλες χώρες να μπουν στην ομάδα, ε, την Ουρουάη ας πούμε, την Ινδία, οι αραβικές χώρες που μπορεί να έρθουν και εκείνες αν έρθει και η Κίνα. Η BRICS, Βραζιλία, Ινδία και η Ρωσία δεν είναι στην ΤΙΣΑ, ούτε χώρες του ΑΣΕΑΝ είναι στην ΤΙΣΑ και θα θέλαμε αυτό να γίνει για να έχουμε αυξημένη πρόσβαση στην αγορά των χώρων αυτών. Η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι καλό που ξεκινήσαν οι διαπραγματεύσεις, αλλά τώρα πρέπει να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν με την Μαλαισία, με το Βιετνάμ, με την Ταϊλάνδη. Όλες αυτές οι χώρες ΑΣΕΑΝ έχουν υψηλές φραγμούς για την πρόσβαση στην αγορά και θα θέλαμε εκεί να σημειωθεί πρόοδος. Η Ινδονησία έρχεται, δεν έρχεται, θέλει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και να επανέλθει αργότερα. Θα θέλαμε η Ινδονησία να μπει στις διαπραγματεύσεις με την Ένωση γιατί είναι ο τέταρτος πληθυσμός στον κόσμο με 240-50 εκατομμύρια κατοίκους. Πολλά υποσχόμενη χώρα κατά τη γνώμη μου. Έπειτα, τι και η Ιαπωνία. Μεγάλη ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. και εστιάζουμε την προσοχή. Υπάρχουν πολλές υποσχέσεις δηλαδή, αλλά πρέπει όλα αυτά να συγκεκριμενοποιηθούν. Τα βάλαμε όμως στη λίγο στην άκρη γιατί οι εταίροι μας δεν ήθελαν να κάνουν κάτι και να πετύχουν κάτι και αλλά ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με την Ινδία, με τη Μερκοσούρ. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η δύο εταίροι, δυστυχώς δεν προχωρούν για την ώρα, αλλά ελπίζουμε πως στο μέλλον θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αναφέρθηκε και η EPA. Είμαστε απογοητευμένοι με το γεγονός γιατί οι συμφωνίες ευρωπαϊκής εταιρικής, οι ευρωπαϊκές συμφωνίες εταιρικής σχέσης δεν ε, αγγίζουν καθόλου τις υπηρεσίες. Και αυτό βοηθά τις χώρες να μην δεσμευθούν για τις υπηρεσίες. Γιατί αν δεν δεσμευθούν αυτές οι χώρες για τις υπηρεσίες δεν πρόκειται να αναπτυχθούν σοβαρά. Τέλος, πολλά από τα στοιχεία της εμπορικής πολιτικής μπορούν να βελτιωθούν. Νομίζω πως η Κομισιόν θα πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία των εισαγωγών. Έχουμε τονίσει πολύ τις εξαγωγές και τις δυνατότητες των χωρών να πουλάνε πράγματα, αλλά χρειάζεται πάντα να έχουμε και περισσότερες επιλογές και αγαθά για τους ε, καταναλωτές και, με, και πιο, πιο, προσιτά. Ξέρω πως η Κομισιόν κάνει κάποια από αυτά και χρειάζεται κάποια ισορροπία εδώ, αλλά ίσως ε, το μήνυμα για το, κίνημα και το, για το Κοινοβούλιο και για τα κράτη-μέλη είναι να είναι αυτό. Εν γέννη για τις διαπραγματεύσεις, για τις ελεύθερες συναλλαγές, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι το εμπόριο, είναι η business και η Κομισιόν έχει βρει μια καλή ισορροπία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και τις ρυθμιστικές πτυχές των διαπραγματεύσεων, αλλά δίνεται έμφαση από τα κρατημέλη και το σώμα αυτό να εστιάσουν σε μη εμπορικά θέματα που ευχαρίστως να είναι μέσα στις συμφωνίες, ας πούμε βιωσιμότητα, εργατικά ε, θέματα ή θέματα περιβάλλοντος. Αλλά τελικά πρέπει να θυμόμαστε πάντα πως αυτές οι συμφωνίες είναι βασικά εμπορικές συμφωνίες. Μια άλλη ιδέα θα ήταν περισσότερα κονδύλια για την γάμα δέλτα εμπορίου. Ε, στην επόμενη επιτροπή δηλαδή θα πρέπει να εστιάσουμε στη σαφήνεια για την ευρωπαϊκή οικονομία και, για, και όπως είπε και ο Γενικός ε, Διευθυντής η ανάπτυξη είναι εκτός Ένωσης. Περισσότερα κονδύλια λοιπόν για την γάμα δέλτα εμπορίου αλλά και για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών. Περισσότερη ίσως διαφάνεια. Θα έλεγα περισσότερες στατιστικές για το εμπόριο στις ε, υπηρεσίες και το FDI. Ξέρουμε ας πούμε πόσα μπουκάλια εισάγονται ή εξάγονται από την Ένωση, αλλά δεν ξέρουμε πολλά για το εμπόριο στις υπηρεσίες εν γέννη και αυτό πρέπει πιστεύω να βελτιωθεί. Τέλος, ίσως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια ε, στην πρόθεση του εμπορίου, διότι νομίζω πως η Κομισιόν και στις Βρυξέλλες το βλέπουμε εδώ, αλλά στα κράτη-μέλη είναι λίγο πιο δύσκολο. Τελευταία μου παρατήρηση, Πρόεδρε, όντως σε κάποιους τομείς των υπηρεσιών έχουμε κάποια αμυντικά θέματα. Ας πούμε τα οπτικοακουστικά είναι ένα, αλλά και στις υπηρεσίες, στις κατασκευές, στις κατασκευαστικές εταιρείες ζητούν ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν για αμοιβαιότητα σε ορισμένα θέματα δημοσίων συμβάσεων είναι κάτι χρήσιμο. Και επίσης η χρήση του αντι dumping και υπηρεσίας στον τομέα αυτό αναφέρθηκε. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και εγώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χέντριξ, που είναι Διευθυντής Πολιτικής για... της, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Βιοτεχνιών. Δεδομένων στη ε, σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα σας ακούσουμε μεγάλη προσοχή κύριε Χέντριξ. Έχετε το λόγο. Πού είστε? Α, μάλιστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, για την πρόσκληση. Όπως είπατε η Ένωσή μας ε, εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και σίγουρα είναι σημαντικές γιατί είναι το 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε την φιλοδοξία να προβούμε σε μια πλήρη αξιολόγηση της ε, θητείας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και των επιδόσεων της σε θέματα εμπορίου, εμπορικής πολιτικής. Είναι εντυπωσιακή βέβαια η δράση της Κομισιόν και το θεματολόγιο στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να κάνω μόνο μερικά γενικά σχόλια για την εμπορική πολιτική. Και ένα από τα πρώτα σχόλια που θέλω να κάνω και νομίζω ότι και ο διευθυντής της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριο, ο κύριος Ντεμαρτή, ε, θα ενδιαφέρεται γι' αυτό, είναι ο τρόπος ε, επικοινωνίας με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριο και πώς και η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριο επικοινωνεί με τους διαφόρους ενδιαφερομένους φόρους. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλές ε, και υπήρξαν πολλές δυνατότητες κατά το παρελθόν να έχει κανείς επικοινωνία με τη ΓΑΜΑ Εμπόριο. Επικοινωνία όμω μεταξύ ε, των εμπλεκομένων φορέων όλων αυτών των φορέων και τη ΔΕΛΤΑ εμπόριο πρέπει να και μπορεί να βελτιωθεί. Περισσότερη διαφάνεια συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων είναι κάτι απαραίτητο και ιδίω για το μέλλον, διότι νομίζουμε ότι ένα από του λόγου τη αποτυχία τη ΑΚΤΑ ήταν ακριβώ το γεγονό ότι δεν ε, υπήρχε διαφάνεια και σε ό,τι αφορά τη συμφωνία IP, ούτε και αυτή θα θέλαμε να αποτύχει, γι' αυτό και επιμένουμε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, για να δώσω ένα παράδειγμα, προθεσμίες για την ε, διατύπωση σχολείων. Πολλές φορές οι προθεσμίες είναι σύντομες, ιδίως για πολύπλοκα θέματα όπως είναι επενδύσεις και υπηρεσίες. Και η επικοινωνία μεταξύ κομισιών και εμπλεκομένων φορέων θα βελτιωθεί εάν οι προθεσμίες ανταποκρίνονται καλύτερα στα αιτήματα και αν υπάρχει και περισσότερη διαφάνεια. Μάλλον υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια. Εμπορικέ πολιτικέ. Μπορείτε να πείτε βέβαια ότι και οι δικές μας οργανώσεις έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Οι εμπορικέ πολιτικές πρέπει να μεταφέρονται ε, πιο ξεκάθαρα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, Το ανέφερε και ο προλαλής σας να μην δίνουμε έμφαση μόνο στις εξαγωγές αλλά και στις εισαγωγές. Διότι συχνά ξεχνιέται ο συνολικός αντίκτυπος των εμπορικών πολιτικών στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ο αντίκτυπος αυτός δεν είναι πάντοτε γνωστός και είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς μια ιδέα ή τέλο πάντων να παρακολουθεί το θεματολόγιο της Κομισιόν στα θέματα του εμπορίου δεν έχει τι απαιτούμενες γνώσεις. Οι πολιτικές λοιπόν θα πρέπει να ε, μεταδίδονται καλύτερα και στις ΜΜΕ. Διότι πολλές από αυτές είναι πολύ αφηρημένες και απομακρυσμένες. Δεν φτάνουν δηλαδή επί τόπου ε, της ΜΜΕ, ούτε και τις οργανώσεις τους. Η διαφάνεια τώρα, η διαφάνεια θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη αποδοχή των εμπορικών πολιτικών της Ένωσης ε, γενικώ από τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και νομίζω και από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες υπάρχουν ε, σημαντικά θέματα όπως είναι η προστασία των επενδύσεων, ε, το ISDS και είναι καλό που συντάσσονται ενημερωτικά δελτία, fact sheets. Τώρα έρχομαι στην εμπορική άμυνα που είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο και λεπτό. Εξού και έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία ε, η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για τον εξυγχρονισμό των μηχανισμών εμπορικής άμυνας. Είναι μια πρόταση λοιπόν ε, που την καλωσορίζουμε αυτή για την επανεξέταση του μηχανισμού, των μηχανισμών εμπορικής άμυνας και ιδίως για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών Αυτά αναφέρονται στην ε, ανακοίνωση της Κομισιόν και είναι πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις ΜΜΕ. Αυτές οι πτυχές πράγματι είναι κρίσιμες ε, για τις επιχειρήσεις. Η έλλειψη πληροφορίων και ε, προβλεψιμότητας μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές και άλλες επιπτώσεις σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Και ιδίω βέβαια αν αυτή είναι μικρομεσαία. Τα μέσα εμπορική άμυνα θα πρέπει να είναι πιο επιχειρησιακά εν γέννη, δηλαδή να τιμωρούν, να κολλάζουν αξιόπινε ε, ε, πράξει ή πράξει που οδηγούν σε dumping. Η αναθεώρηση των προθεσμιών είναι σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση, αλλά τα χρονοδιαγράμματα ορισμένε φορές είναι πολύ ανεδαφικά και περιορισμένα χρονικά. Θα πρέπει Επίσης η διαδικασία να διευκολύνει το δυνατόν περισσότερο και αν όχι να χρησιμοποιούνται ε, φιλικά προς το χρήστη εργαλεία και να υπάρχουν και εγχειρίδια που τους μη μονομαθείς να τους καθοδηγούν σε ό,τι αφορά τα έγγραφα και τα ερωτηματολόγια που θα πρέπει να καταρτίζουν. Επίσης, δημοσιοποίηση και κατάρτιση κατευθυντηρίων γραφών, γραμμών τη βελτίωση της ε, διαφάνειας και της προβλεψιμότητας σε διάφορους τομείς για να μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιολογούν καλύτερα την κατάστασή τους. Επίσης, αναβάθμιση του help desk και ε, αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους, γιατί αυτά τα help desk ε, πολλές φορές βοηθούν πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποφεύγουν έτσι τις υψηλές αμοιβέ ε, για νομικές υπηρεσίες, νομικών υπηρεσιών. Τώρα, για τις δραστηριότητες στην ΚΑΜΑΔΕΛΤΑ εμπόριο. Θέλω να μιλήσω για τη διεθνοποίηση πολλών ΜΜΕ. Μέχρι το 2015 το... Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ίσως το 90% θα ε, γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα έχουμε το επίπεδο του 43%. Όταν λέω διεθνές εννοώ εξαγωγές και εισαγωγές. Είναι σημαντικό λοιπόν το να βγουν προς τα έξω οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να γίνουν προσπάθειες και σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Πού μπορεί λοιπόν να προσφέρει προστέμενη αξία, ε, σε ποιους τομείς η Ευρώπη. Για παράδειγμα, εμπορική πολιτική πρόσβαση στις αγορές, και βάση δεδομένων σχετική άσκηση πιέσεων με ευρωπαϊκή διάσταση, πληρωματικά προγράμματα σε περίπτωση στοχιών των αγορών, εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ. και μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική για την παροχή τυποποιημένων πληροφοριών σε στοχευμένες αγορές τρίτων χωρών. Είναι κάτι που πραγματικά ε, το περιμένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερη ορατότητα των υφιστάμενων μηχανισμών στήριξης των ΜΜΕ και των σχετικών δομών. Αυτά θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ε, υπηρεσιών. Η διεθνοποίηση λοιπόν, αυτή η διαδικασία για να είναι επιτυχημένη χρειάζεται στήριξη και σε τοπικό επίπεδο όχι μόνο στο εξωτερικό. Αυτή η προσέγγιση δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ε, στις ε, πρωτοβουλίες της Κομισιόν μέχρι τώρα. Στο μεγαλύτερο τμήμα του δαπανάται σε δομές σε τρίτες χώρες και σε υπηρεσίες που παρέχονται και οι υπηρεσίε που παρέχονται σε επίπεδο κρατών μιλών θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ΠΟΕ, χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα του Μπαλί και οι διαπραγματεύσει πιστεύουν ότι θα πρέπει βέβαια να συνεχιστούν. Η πολιτική τη ε, Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ ε, θεωρούμε ότι είναι θετική. Θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία σύναψη συμφωνιών με τρίτε χώρε και θα πρέπει να οδηγήσουν οι σχετικέ συμφωνίε σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση για να ωφεληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό. Επίση, θα προτιμούσαμε και εμεί την πολυμερή προσέγγιση Βέβαια, οι διμερείς επαφές ε, είναι και αυτές ε, θεμητό μέσο η προστασία των δικαιωμάτων πραγματικής ε, ιδιοκτησίας στις νέες συμφωνίες ε, είναι σχεδόν μια τυποποιημένη διαδικασία και το θεωρούμε θετικό. Θα πρέπει να συνεχίσει την προσέγγιση αυτή η Κομισιόν, θα πρέπει να συνεχίσει να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα σε όλες τις μελλοντικέ συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Και επειδή οι δύο ΜΜΕ έχουν προβλήματα στο να ε, περασπιστούν γενικώ τα πνευματικά δικαιώματα, ιδίω σε διεθνέ πλαίσια. Τέλο, η αρχή τη αμοιβαιότητα πρέπει να ε, εδρεωθεί, να υπάρχει δηλαδή ένα νομικά δεσμευτικό εργαλείο που θα συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέσα ελέγχου για να έχουμε ένα θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπορικών τη εταίρων. Θετική είναι επίση και η εστίαση στη μείωση των μη δασμολογικών φράγμων στι διαπραγματεύσει συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Τελευταία λέξη για το πρόγραμμα TTIP. Το χαιρετίζουμε φυσικά, αλλά ε, πρέπει να πω ότι περιμένουμε και μεγαλύτερη απασχόληση και ανάπτυξη χάρη σε αυτή τη συμφωνία. Και περισσότερο από, ότι από άλλες ε, συμφωνίες εμπορίου λόγω των στενών δεσμών μεταξύ των δύο συμβαλωμένων πλευρών. Περιμένουμε να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια, συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων. Τα βλέπουμε αυτά. Λέμε ότι στη συμβουλευτική ομάδα που συγκρότησε η Κομισιόν έχει υπάρξει κάποιο σφάλμα ε, σε σχέση με την ε, σύνθεση δεν υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση όλων των πλευρών. Ιδίω ό,τι αφορά τι ΜΜΕ. Νομίζω ένα εκπρόσωπο υπάρχει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν ξεπέρασα το χρόνο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει ο κύριος Σουκούπ. Εμπειρογνώμων. της ε, Αυστριακής οργάνωσης εργασίας. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλες και όλους κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο Μορέιρα για την πρόσκληση που απίφθινε στην Αυστριακή, στο Αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας για να ε, μπορέσει να συμμετάσχει στη συζήτηση. Πρώτα, οι στόχοι τους οποίους θα πρέπει να επιδιώκει η εμπορική και επενδυτική πολιτική της Ένωσης πριν να προχωρήσω σε κάποια πιο οριζόντια θέματα. Η κοινή εμπορική πολιτική βασίζεται στους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Το άρθρο 3 παραγραφός 5 της ε, Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει τους στόχους, για παράδειγμα μεταξύ άλλων βιώσιμη ανάπτυξη, αλληλεγγύη και αμοιβαίωση σεβασμό μεταξύ των λαών, ελεύθερο και έντιμο εμπόριο, εξάλληψη της φτώχειας και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στα πλαίσια της αξιολόγησης που διεξάγουμε σήμερα είναι σημαντικό να εξεταστεί και η συνοχή της πολιτικής, αν όντως δηλαδή η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όντως εξυπηρετεί τους στόχους που ανέφερα στην πράξη. Η εμπορική και επενδυτική πολιτική της Ένωσης στοχεύει και σε θέματα πέραν των συνόρων και ορισμένοι λένε ότι μπορούμε με το εμπόριο να ξεπεράσουμε την κρίση. Αυτά λέει και στην ανακοίνωσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι παραπλανητικό. 88% της τελικής ζήτησης προσφοράς υπηρεσιών και αγαθών προκύπτει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η εγχώρια ζήτηση μέσα στην ενιαία αγορά είναι πολύ πιο αποφασιστική για την ε, ανάπτυξη της Ένωσης και αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Δοθέντων των στόχων πολιτικής και της ε, ισχύω της ενιαίας αγοράς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και την ευθύνη και την ικανότητα να αλλάξει τις πολιτικές, να ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση στην Ένωση και να λάβει υπόψη και την ανάγκη δίκαιας κατανομής. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, βλέπετε και στο γράφημα ότι υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη μετακίνηση προς την κατεύθυνση των διμερών FTA και αυτό το βλέπουμε εμείς με κάποια ανησυχία διότι θεωρούμε ότι ο αριθμός των διμερών ε, συμφωνιών έχει ε, το δυναμικό να υπονομεύσει την ισχύ των πολυμερών συμφωνιών. Είδαμε την θετική εξέλιξη στο Μπαλί, αλλά δεν νομίζουμε ακόμη ότι υπάρχει αναβίωση των πολυμερών συμφωνιών, διότι ακόμα οποιαδήποτε συμβιβασμή είναι μακριά. Σας υπενθυμίζω βεβαίως το, τη σημασία του πολυμερούς επίπεδου. Τώρα ορισμένα κέρια οριζόντια θέματα που θα ήθελα να σας εξηγήσω σε σχέση με την ποικιλία των συμφωνιών της Ένωσης και ξεκινώντας από τις προδιαγραφές εργασίας της Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Ελευθερών Συναλλαγών Υπάρχουν οι σχετικές διατάξεις, όμως έχουν ορισμένα σημαντικά, ορισμένες σημαντικές ελλείψεις. Η πιο σημαντική έλλειψη για την βιωσιμότητα είναι ότι δεν είναι δεσμευτικές, δεν είναι εξαναγκαστές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες. Εφόσον παραβιαστούν, οδηγούν μοναχά σε κυβερνητικές διαβουλεύσεις ή μη δεσμευτικές ε, συμβουλές ε, ειδημόνων. Γι' αυτό προτείνουμε εμείς, αλλά και απαιτούμε, ο σχετικός μηχανισμός να είναι εξαναγκαστός και συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ε, προδιαγραφών εργασίας να οδηγεί στην επιβολή προστήμων. Επίσης, για τα κεφάλαια βιωσιμότητας θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις για να εφαρμόζονται στο νόμο και στην πράξη όλα, όλες οι προδιαγραφές του, οργανισμού, του Διεθνούς Μάλλον Οργάνωσης Εργασίας. Πάντως, όταν εξετάζουμε την ε, Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέας, δεν περιλαμβάνει παρά μόνο μια αδύναμη ρήτρα ότι θα πρέπει να γίνουν διαρκείς προσπάθειες για να ενισχυθούν οι συνθήκες του, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που δεν έχει ακόμα υπογράψει η Νότια Κορέα. Ιδιαίτερα προβληματικό, από την, ε, προβληματική μάλλον, είναι η FTA με Περού και Κολομβία, όπου εκεί υπονομεύεται η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων διότι λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες των χωρών. Και επειδή η Κολομβία είναι η πλέον επικίνδυνη χώρα για τους συνδικαλιστές, η Αυστρία ζήτησε την μη κύρωση της σχετικής συμφωνίας. Σημειώνω επίσης τη σημασία των ε, βημάτων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών, πολύ σημαντικών για την διατήρηση του διαλόγου μεταξύ κοινωνικών εταίρων, μη κρατικών οργανισμών και των αξιωματούχων των μερών, των συμβαλωμένων μερών στις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Επίσης έχουμε προτείνει οι κυβερνήσεις να είναι υποχρεωμένες να αντιδρούν σε καταγγελίες των ε, συνδικαλιστών. Άλλη μεγάλη ανησυχία για μας είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προστασία των επενδύσεων. Στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να επιτρέψουν σε διεθνείς εταιρείε να προσφύγουν σε διεθνή διαιτητικά δικαστήρια για να προσβάλλουν δημοκρατικές αποφάσεις κυβερνήσεων Ιδίω όταν βλέπουν ότι κινδυνεύουν τα κέρδη τους. Και ιδίω όταν τέτοιοι ισχυρισμοί, όπως γνωρίζουμε, μπορούν να υπονομεύσουν σοβαρά εθνικές πολιτικές εθνική δημοκρατική κυριαρχία αλλά και από την νομική σκοπιά υπονομεύουν το διεθνές νομικό σύστημα και οδηγούν σε διάκριση σε βάρος των εγχώριων επενδυτών. Σε αυτές τις υποθέσεις ISDS είναι πιο προβληματικό ακόμη διότι τα διαιτητικά δικαστήρια που προανέφερα στην ουσία αποφασίζουν και κλεισμένων των θυρών συχνά για την μοίρα μεγάλων ποσών από τα χρήματα των φορολογουμένων. Και είναι προβληματικό διότι δεν υπάρχει και δυνατότητα να εφεσιβληθούν οι αποφάσεις αυτές. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές απειλές. Το 2009 η σουηδική εταιρεία Vattenfall ζήτησε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στη βάση διμερού συμφωνίας από τη γερμανική κυβέρνηση λόγω περιβαλλοντικών προτύπων για ένα σταθμό παραγωγής ρεύματος από άνθρακα. Το 2012 η ίδια Βάτενφαλ προσέφηκε κατά της Γερμανίας. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι και μεγάλες βιομηχανικές ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν παρόμοιες απειλές. Ενώ παλαιότερα νομίζαμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μονάχα στην περίπτωση αναπτυσσομένων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση για το θέμα των επενδύσεων. Νομίζομαι όμως ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι επαρκής, διότι παρόμοιες διατάξεις προβλέπονται και για άλλες ε, συμβάσεις για τις συμφωνίες ΣΥΤΑ για παράδειγμα, όπου δεν γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις, ΣΕΤΑ δηλαδή. Άλλο θέμα τώρα, επίσης σημαντικό για μας, η διασφάλιση των δημοσίων υπηρεσιών. Για μας οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να παραμείνουν εκτός των συμφωνιών αυτών. Το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό πρέπει να διευκρινιστεί τι σημαίνει δημόσια υπηρεσία στο τοπικό και εθνικό επίπεδο και πώς ρυθμίζονται. Η Κομισιόν προχωρεί τώρα σε επιθετικές προσεγγίσεις με συμφωνίες απελευθέρωσης δημοσίων υπηρεσιών. Και αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι η συμφωνία TTIP περιλαμβάνει αρνητική λίστα. Ακολουθεί δηλαδή την ε, προσέγγιση list it or lose it. Και αυτό αποτελεί τη βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσει. Επίσης, να σημειώσω ότι η πρόσφατη πρωτοβουλία πολιτών δικαίωμα στην παροχή νερού δείχνει την ανάγκη προστασίας των δημόσιων υπηρεσιών, των δημοσίων κοινοφελών οργανισμών ή υπηρεσιών. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι παραχωρήσεις για την προσφορά δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να μείνουν εκτός εμπορικών συμφωνιών. Τέλος, θέλω να έρθω σε θέματα διαφάνειας. Δεν νομίζω ότι η εμπορική πολιτική κυρίως αφορά τις επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι μια ποικιλία τομέων επηρεάζεται από τις πολιτικές αυτές. Θεωρούμε ότι για να μπορούν να βασίζονται οι δημοκρατικά λαμβανόμενες αποφάσεις σε νομιμότητα στον δημόσιο τομέα δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε μυστικότητα στη λήψη τους. Και γι' αυτό προτείνουμε οι εντολές και τα έγγραφα για τις διαπραγματεύσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν προσιτά στο κοινό για δημόσια συζήτηση, να γίνονται πραγματικές διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να περιληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει δηλαδή σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νομίζουμε ότι αυτά τα συμπεράσματα είναι σημαντικά για να μπορέσουν να βασιστούν οι εμπορικές πολιτικές σε μεγαλύτερη βάση νομιμότητας. Σας, Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια. Η κυρία Ούλμεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Είμαι και μέλος της ε, Concourse. Προσπαθώ να μιλήσω εξ ονόματος ε, της ε, Concord επίσης, εκτός από την Απροτεύ. Έχουν υπάρξει διάφορες εξέλιξεις τα τελευταία 5-6 χρόνια. Η ομιλήτρια χωρίς μικρόφωνο. I would think that most of the amendments of the οι περισσότερες αλλαγές, ε, που, μάλλον τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι ΜΚΟ που ασχολούνται με την ανάπτυξη, δεν έχουν ληφθεί υπόψη ε, στις, ε, στην νομοθεσία. Αυτή είναι μια πρώτη γενική παρατήρηση. Θα σας μιλήσω για την αναπτυξιακή πολιτική και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εμπορικές πολιτικές, τις επενδύσεις και κάποιες συστάσεις. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας αυτό που είδαμε είναι ότι η Ένωση ε, με την εμπορική της πολιτική ηγείται του σχηματισμού της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής γιατί η εξωτερική της πολιτική είναι σχετικά δύναμη και δεν είναι αρκετά συνεκτική ανάμεσα στα κρατημέλη και αυτό μας ανησυχεί. Ακούμε ότι η ατζέντα αυξάνεται, ε, παίρνει τεράστιες διαστάσεις και κατά κάποιο τρόπο σχηματίζει τις κατευθύνσεις για την εμπορική πολιτική. Ανησυχούμε πολύ για την ποιότητα της ανάπτυξης και όχι μόνο για την ποσότητα. Αναφέρθηκε και από την πλευρά των συνδικάτων ότι η ανάπτυξη του ΕΠ δεν μεταφράζεται αυτόματα σε οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό δεν το έχουμε ακούσει και πολύ τα τελευταία χρόνια από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Όταν, όσον αφορά τον ΠΟΕ, τις διμερείς, πολυμερείς ε, διαπραγματεύσεις, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά δεν επιτρέπει όλες, όλες τις χώρες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα διάφορα στρώματα. Ας πούμε, ένα παράδειγμα, είδατε την προσφορά για τις επιστροφές στις εξαγωγές στην γεωργική πολιτική. Ο Επίτροπος Τσόλος το έχει προσφέρει αυτό σε ένα είδος ε, ε, επιθετικής ε, έλκυση των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα επίπεδα διμερείς ή πολυμερείς ε, διαπραγματεύσεις και το κάνει σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα, αλλά βάζει σε πολύ αδύναμη θέση πολλές άλλες χώρες. Σε σχέση με τα ε, κεφάλαια της βιωσιμότητας Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει εκεί δυνατότητα επιβολής και θα είναι πρόκληση να συμμετέχουμε σημαντικά στα κεφάλαια της βιωσιμότητας επειδή είναι σχετικά μικρά τμήματα των διαφόρων ε, συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Αναπτυξιακή πολιτική και σύγκρουση ανάμεσα στο εμπόριο και την ανάπτυξη πιστεύουμε πως δεν έχουν νόημα όλα αυτά ε, μέσα στην εμπορική πολιτική της Ένωσης. Το εμπόριο μπορεί να είναι προοδευτικό ή να είναι οπισθοδρομικό, αλλά εξαρτάται από τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς και ότι η βέλτιστη κατανομή της παραγωγής δεν γίνεται απαραίτητα μέσω του ελευθέρου εμπορίου και των σχετικών συμφωνιών. Ωστόσο, η κατανομή αφήνεται στις εγχώριες πολιτικές και δεν μπορεί αυτό να ανατίθεται στις εγχώριες πολιτικές. Θα πρέπει να καταλάβουμε πώς επηρεάζει το εμπόριο, τα κοινωνικά και άλλα συμφέροντα στις χώρες αυτές, γιατί ξέρουμε πως το εμπόριο δημιουργεί, μπορεί να δημιουργήσει και δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και γι' αυτό και θα πρέπει η Ένωση να ασχοληθεί με το πώς η απελευθέρωση του εμπορίου και η ανάπτυξη του εμπορίου επηρεάζουν τις υπόλοιπες πτυχές. Αυτό δεν λαμβάνεται αρκετά υπόψη στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Τώρα, όσον αφορά Ορισμένες εμπορικές πρωτοβουλίες, ορισμένοι από εμά παρακολουθήσαμε την ακρόαση ΕΠΑ εδώ στο Κοινοβούλιο, σε αυτή την Επιτροπή και η αξιολόγηση είναι ανάμεικτη. Είδαμε ότι ορισμένες χώρες έχουν υπογράψει το, για το εμπόριο γιατί λάβαν βοήθεια, δηλαδή είναι το εμπόριο ένα άνοιγμα για τη βοήθεια. Δεν είναι ένα αντάλλαγμα. Θεωρείται δε Ε, ότι πολλές χώρες έχουν λάβει βοήθεια ε, ώστε να ανοίξουν ε, τις αγορές, τις, για το, τις αγορές τους για το εμπόριο. Υπάρχουν αμφιβολίες λοιπόν για το πώς γίνεται αντιληπτή η Ευρώπη σε όλες αυτές τις χώρες. Τώρα το, για το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων, ορισμένες, πολλές μάλλον οργανώσεις αναπτυξιακές προτι, προσπαθούν να προτείνουν περισσότερους δείκτες εκτός από το ΑΕΠ, να, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή δείκτες που είναι φιλικοί προς την ανάπτυξη για να έχουμε διαφορετικά ε, αποτελέσματα όπως οι δείκτες της οικονομικής ε, ευαισθησίας ή των ανθρωπίνων πόρων. Το γεγονός ότι έχει μεταρρυθμιστεί το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων δεν σημαίνει ότι αφήνει χώρο ε, επιλογής για τις χώρες που δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Και αυτό μας λυπεί. Τώρα, όσον αφορά τι εμπορικέ πολιτικέ και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει, πιστεύουμε, σύγκρουση ανάμεσα στην εμπορική νομοθεσία και το διεθνές ε, δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δικαίωμα ε, τροφή και πολλές ε, ε, ε, εκθέσεις του ΟΗΕ από τον ειδικό εντεταλμένο για τη διατροφή, τον κύριο Ντεσελιέ, βλέπουμε ότι το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες δεν προβλέπουν δεν, είναι συμβατές μάλλον και, οι κανόνες του ΠΟΕ εμποδίζουν και καθορίζουν την ε, διατροφική πολιτική για πολλές χώρες. Το αποτελέσμα, το πούμε, στην Ινδία είναι χαρακτηριστικά ε, και κραυγαλαία για αυτό το σύστημα και την ασφάλεια των τροφίμων. Πιστεύουμε πως ε, πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση για το πώς το διεθνές εμπορικό δίκαιο αλλά και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρωπίνα δικαιώματα συνδυάζονται και τι ε, κυριαρχεί τελικά. Τώρα, έχουμε και το θέμα της ε, Καμπότζης. Ε, θεωρούμε πως είναι ένα αποτέλεσμα των των, των μεταρρυθμίσεων που έγιναν είχαμε μέσα τη μεταρρύθμισης του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων μια όθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετά από τέσσερα χρόνια υποβολής αιτήσεων Πολλές ε, οργανώσεις ή ενώσεις ε, που είναι ε, στην Καμπότζη δίνουν αποδείξεις για παραβιάσεις, αλλά δεν θα πρέπει μόνο η Κομισιόν να αποφασίσει αν θα ενεργοποιηθεί μια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λυπούμεθα που τελικά η μεταρρύθμιση δεν έχει οδηγήσει σε αποτελέσματα. Επίσης πιστεύουμε πως ίσως οι διαπραγματεύσεις TTIP θα, θα φέρουν κάποιες από αυτές τις συζητήσεις για την συνοχή ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ε, ξανά στο επίκεντρο και θα κινητοποιήσουν ε, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς γιατί πιστεύουμε πως η ατζέντα αυτή θα επηρεάσει ένα μέγα φάσμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και στις ευρωπαϊκές χώρες και ως προς αυτό μπορεί να κινητοποιήσει την προσοχή. Όσον αφορά τις ε, αρμοδιότητες της Ένωσης για τις επενδύσεις, εξακολουθούμε να ακούμε τις ίδιες δηλώσεις, ότι δηλαδή οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι καλές και οθούν την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη οδηγεί σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά τι είδος ανάπτυξη και τι είδος θέσεις απασχόλησης λέμε εδώ. Εμείς ε, βλέπουμε αντίθετα ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις δίνουν κέρδη στις εταιρείες, αλλά δεν σέβονται απαραίτητα ή δεν προωθούν απαραίτητα την ε, κοινωνική ή περιβαλλοντική ανάπτυξη. Τώρα, τι είδαμε στη Μιανμάρ, ήμασταν ε, εμείς ε, φυλακτικοί όσον αφορά την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ε, Μιανμάρ, αλλά υπάρχει μια τάση για κέρδος. Δεν οθούνται όλα, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις από ανθρωπιστικές ή περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλά από το κέρδος Τώρα, για τη διαφάνεια, το αίτημα είναι σαφώς ε, να είναι τα κείμενα ανοιχτά και προσιτά, γιατί διαφορετικά υπάρχει χάσμα στη διαφάνεια, δεδομένου ότι αυτές οι διατάξεις θα επηρεάσουν πολλές, πολλές πτυχές καθημερινής ζωής. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή ΙΝΤΑ, είδαμε υπάρχει το δίλημα της αυξανόμενης ε, σημασίας της ε, συναπόφασης για το Κοινοβούλιο, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σε πολλές, σε περισσότερες ε, συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών, με αποκλεισμό δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή για να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς κάποια από τα εμπιστευτικά κείμενα, γιατί αυτά που είναι εμπιστευτικά σημαίνει πως αυτοί που, που είναι οι πιο ισχυροί μάλλον θα δουν τα κείμενα ενώ το ευρύ κοινό δεν ε, παίρνει είδηση τι συμβαίνει. Θα θέλαμε επίσης να έχουμε και την ε, επικοινωνιακή πολιτική της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου να εντοπίζει και στις κινδύνους και στις απώλειες και να μην αναφέρεται μόνο στις περιστάσεις ε, win-win γιατί από την εμπειρία μας υπάρχουν πάντα οι χαμένοι. Τώρα, όσον αφορά τις συστάσεις, έχω ήδη αναφέρει κάποιες, ίσως ακόμα μία. Ο νέος ειδικός συζητητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Σταύρος Ραμπρινίδης έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις και θα θέλαμε να δούμε απάντηση από το επόμενο κοινοβούλιο και από την Κομισιόν. Επίσης λέει ότι υπάρχει μια έκθεση στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Παρακαλώ κλείστε. Και θα θέλαμε να δούμε λοιπόν θετική ανταπόκριση από την Επιτροπή σας σε αυτές τις συστάσεις και σας ευχαριστώ. Um... Πριν ε, ξαναδώσω τώρα στον κύριο Ντεμαρτή, να κάνω κάποια σχόλια. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής μας θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την ε, επικοινωνία μας προς τα έξω και προς τα εσάς ε, δεν υπάρχει άλλος μετά από μας. Ποιος οργανώνει τέτοιες ακροάσεις. Ε, διαρωτώ με. Υπάρχει άλλος που μπορεί ε, να πει κάποια άλλη επιτροπή ε, εμπορική, κάποια άλλο θεσμό τέτοιο που να πει ότι έχει περισσότερη διαφάνεια. Ο κύριος Δεμαρτή. Οι βουλευτές δεν θα μιλήσουμε, λέει ο κύριος Ζαντό. Ο πρόεδρος. Νόμιζα ότι ήμουν μόνο μου, γιατί στην αρχή ήμουν μόνος μου, λέει ο πρόεδρος. Ε, εντάξει, να δώσω το λόγο στα μέλη λοιπόν. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Ακούσαμε διαφορετικές αξιολογήσεις της εμπορικής πολιτικής. Ιδίως η τελευταία αξιολόγηση, εκεί πρέπει να γίνει πάλι κάποια διαφοροποίηση σχετικά με το ποιος έχει καταθέσει ποιες θέσεις στην Επιτροπή, η οποία Επιτροπή δεν είναι ον άνευ έχει απαρτίζεται από μέλη τα οποία καταθέτουν προτάσεις και τροπολογίες. Θέματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών εδώ έχουν τεθεί και από τα μέλη, δηλαδή από τους βουλευτές. Πάντως ήθελα να επανέλθω στις EPA. Τις Ευρωπαϊκές συμφωνίες εταιρικής σχέσης που αυτές απετέλεσαν και την βάση για την αξιολόγηση της εμπορικής πολιτικής. Τέτοιες συμφωνίες βρίσκονται στην φάση των διαπραγματεύσεων επάπειρο χρόνο και ακούω ξανά και ξανά ότι επίκειται η ολοκλήρωσή τους και πάλι περνούν δύο-τρία χρόνια. Δεν μπορώ λοιπόν να εκτιμήσω πολύ καθαρά πού εντοπίζεται ο σχετικός προβληματισμός και πού, εν ώψη και των επικρίσεων που ακούσαμε, θα πρέπει να προσπαθήσω να κάνω ένα βήμα προς τα εμπρός, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να προκύψει και κέρδος για τις συμβαλόμενες χώρες, αλλά και για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Ίσως μπορούμε να ακούσουμε τις κριτικές αυτές λοιπόν και να δώσουμε κάποιες εξηγήσει στη βάση του παραδείγματος των EPA. Ευχαριστώ, Μπέρντ, από τους πράσινους, ο σκιώδης συγητής. Κύριο Ζαντό, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καθησυχάσω τους φίλους και εκπροσώπους που ήταν εδώ ότι δεν λέμε τίποτε απόρριτο στις και κλεισμένα των θερών συνεδριάσεις. Συχνά είναι συμπαθητικές, αλλά μην φανταστείτε ότι έρχεται ξαφνικό κύριος Ντεμαρτή και μας ε, ε, αναφέρει και μας εξηγεί το σκληρό πέραν διαπραγματεύσεων, ε, απλά ε, σίγουρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν και κάποιοι χώροι αντιπαράθεσης ίσως με την Κομισιόν και με τις υπηρεσίες, αλλά μην φανταστείτε ότι αν μπει ένας κοριός και ακούσει τι λέμε εδώ θα μάθει όλα τα μυστικά του Κοινοβουλίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ε, ευρωπαϊκή στρατηγική, έχω δύο έντονες επιφυλάξεις. Το πρώτο, εσωτερική συνεκτικότητα και συνέπεια. Έχω ένα πρόβλημα με την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Το είπε και ο κύριος Διευθυντής. Σήμερα η Ευρώπη έχει πολύ φορτωμένο και διαφοροποιημένο θεματολόγιο διαπραγμάτευσης. Η Ευρώπη έχει τα εμπορικά, αμυντικά και επιθετικά συμφέροντα για κάθε ε, διαπραγμάτευση. Έχουμε χαμένους, έχουμε κερδισμένους. Κάποιους τομείς τους αφήνουμε, κάποιους τους περασπιζόμαστε. Αλλά τελικά η ισορροπία σε κάθε διαπραγμάτευση την χάνεται μεταξύ των συμμαχίας αυτών που έχουν ε, επιθετικά συμφέροντα κατά τι συμμαχίε που έχουν αμυντικά συμφέροντα, αλλά ουσιαστικά δεν μα διχάζει κάτι σε ό,τι αφορά ε, τι επιδιώξει μα για την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Το γεγονό όμω ότι δεν έχει βιομηχανική πολιτική η Ευρώπη και το ότι δυσκολεύεται να έχει και μια οικονομική άποψη της ανάπτυξης, ένα οικονομικό όραμα για την ανάπτυξή της, αυτό δημιουργεί πολλές από τις ε, δυσκολίες που αντιλαμβανόμαστε στην Επιτροπή μας και που βλέπουμε. Ε, και τίθεται το ερώτημα τι οικονομία θέλουμε για το μέλλον. Και υπάρχει και έπειτα και το ζήτημα της εξωτερικής συνεκτικότητας ε, και συνέπειας. Υπάρχει μια συζήτηση γύρω κυρίως από τη Διατλαντική Συμφωνία για την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία και ποια είναι η θέση της Ευρώπης ε, στην παγκοσμιοποίηση η ισορροπημένη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας, ήπα αναδυόμενων χωρών. Και η συζήτηση αυτή και στη δική μας Επιτροπή δεν νομίζω ότι έχει διεξαχθεί σε επαρκή βαθμό και δεν το λένε μόνο οι πράσινοι. Διαβάζω ένα από τα έγγραφα κάποιου προκατόχου σας, τέλο πάντων, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς, ο κύριο Ντεφρέν για παράδειγμα. Ε, ε για την ισορροπία και ποια είναι η θέση της Ευρώπης στην παγκοσμιοποίηση. Με τη Διατλαντική Συμφωνία, για παράδειγμα, μήπως πάρα πολύ εύκολα μπαίνουμε στη στρατηγική τον είπα για κάποια έτσι, παρεμπόδιση της ε, Κίνας. Σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο ε, χαρακτηριστική ήταν η διέρεση της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τα κινέζικα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ας ε, αφήσουμε κατά μέρος τις ιδιαιτερότητες ε, αυτών των φωτοβολταϊκών συστημάτων από την Κίνα. Τα κράτη-μέλη ήταν πάρα πολύ διαιρεμένα και δημοσία μάλιστα. Δεν το λέγανε μόνο στις ε, συνεδριάσεις γιατί αυτό θα ήταν κατά κάποιο τρόπο και φυσιολογικό να υπάρχουν αποκλήσεις. Αλλά και στη σκηνή τη, τη δημόσια ήταν πολύ διαιρεμένη η Κίνα εποφελήθηκε από αυτή την ε, δημόσια απόκληση απόψε μεταξύ των Ευρωπαίων. Αυτή την έλλειψη συνεκτικότητας και ενότητας της Ευρώπης απέναντι σε ένα τέτοιο εταίρο ε, πρέπει να την προσέξουμε γιατί είναι πολύ επιζήμιο για τα συμφέροντά μας αυτό. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Ντεμαρτή. που έχει να κάνει με το γενικότερο αυτό πλαίσιο. Το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να επικυρώσει αυτό το νέο ε, γενετικό τροποποιημένο οργανισμό, ε, τον αραβόσιτο, είναι κάτι καλό αυτό σε σχέση και με τις διαπραγματεύσει μας ε, με τους Αμερικανούς για το TTIP. Και ένα ερώτημα προς τους φίλους μου για τις υπηρεσίες. Νομίζω και καταλαβαίνω βέβαια ότι οι υπηρεσίε σίγουρα είναι και επιχειρήσεις, ε, business κατά κάποιο τρόπο. Τι θα πούμε, η ε, πρόκειται για επιχείρηση και μη μας ε, αναφέρετε καμία άλλη παράμετρο. Νομίζω ότι στο δικό σας πεδίο παρέμβασης έχετε πάνω χάρη τις υπηρεσίες υδροδότησης. Το να πούμε ότι σήμερα το θέμα της απελευθέρωσης των υπηρεσιών υδροδότησης έχει μόνο οικονομικά διακυβεύματα, ε, νομίζω δεν θα ήταν μια σόφρον προσέγγιση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί το νερό είναι ένα κοινό αγαθό, ένα αγαθό για την ανθρωπότητα. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά αυστηρό στις επιχειρήσεις. Θα ήταν σφάλμα να το θεωρήσουμε έτσι, θα ήταν μια ασφαλμένη προσέγγιση. Τι ερώτημα όμως έχω να σας θέσω Αναφερθήκατε και στη συμφωνία με το Κάρι Φόρουμ, ε, το ε, αυτό το θέμα των φορολογικών παραδείσων, απελευθέρωση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πού το εντάσσουμε αυτό από τη στιγμή που η φοροδιαφυγή και η φορολογική παράδειση και ε, οι χρεώσει των εμβασμάτων κτλ. Ε, είναι ένα θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι πιστεύετε παραδείγματος χάρη για τις δημόσιες συμβάσεις. Σήμερα η Ευρώπη προσπαθεί και μιλάει για την απελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων ε, με θετικό τρόπο. Είπα, το 23% νομίζω των δημόσιων συμβάσεων το έχουν αποκλειστικά για τις δικές τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πως είναι στρατηγικό σφάλμα και εμείς πρέπει να απελευθερώσουμε πλήρως ή θέλατε να έχουμε και εμείς ε, να δώσουμε το ίδιο ακριβώς επίπεδο και ποσοστό προτίμησης ε, στις δικές μας επιχειρήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συνδικάτα. Έθεσα το ερώτημα και το πρωί στην κυρία Σεγκόλ. Δεν έχω καταλάβει αν για παράδειγμα. Νίκα, λέει ο πρόεδρος, ε, δεν υποτίθεται ότι θα απαντήσουν σε ερωτήσεις μας οι προσκεκλημένοι μας. Στην Επιτροπή ε, και εμείς και οι ίδιοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους. <laughs> Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα θέσω το ε, ερώτημα στον Επίτροπο, λέει ο κ. Έχω Έχουμε ένα ερώτημα, επειδή αναφέρθηκε πολύ το θέμα της διαφάνειας. Πώς ε, διαχειρίζεστε αυτό το θέμα που επανέρχεται Μονίμω στις διαπραγματεύσεις, ιδίως με τις εκβιομηχανισμένες χώρε, αλλά όχι μόνο. Είμαστε σε αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της κοινωνίας, την ε, δημοκρατία και ε, ε, φαντάζομαι ότι όπως και εμείς ούτε και εσείς μπορείτε εύκολα να εξηγήσετε σε έναν σκεπτόμενο πολίτη ότι εσείς διαπραγματεύεστε επιλογές της κοινωνίας και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση, είτε πρόκειται για την Ιαπωνία, είτε για τον Καναδά και βέβαια και για τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Uh, finally, Σοπόλ Μέρφυ από την Κούε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη του πάνελ. Υπάρχει ένας ε, χρόνος ε, για τα μέλη ε, για να κάνουν καταληκτικές παρατηρήσεις. Αυτό λέει η μερική άρα θα μπορούσαν ίσως να απαντήσουν. Λοιπόν, αν δούμε τον ε, απολογισμό ε, της ε, δραστηριότητας της Επιτροπής, εξαρτάται αν θα το δεις θετικά ή όχι, το τελικό αποτέλεσμα, το ποια είναι η άποψή σου, αν είσαι νεοφιλελεύθερος, αν είσαι πιο πολύ υπέρ του προστατευσμού κτλ. Υπάρχουν υπέρ και κατά και εξαρτώνται όλα από το πώς θα βλέπει κανείς τα πράγματα. Το υπέρ, το πλεονέκτημα κατά τη δική μου άποψη, ό,τι αφορά τη θητεία της Επιτροπής μας, ήταν ε, η αποτυχία της ΑΚΤΑ που έδειξε ότι αυτές οι εμπορικές πολιτικές ε, όταν εκτεθούν ε, στους προβολείς δημοσιότητας και της κοινή γνώμης καταραίουν εάν υπάρχει κινητοποίηση. Και στην περίπτωση της ΑΚΤΑ αυτό συνέβη. Και φαντάζομαι ότι φοβάται και η Κομισιόν πως συμβεί και αντίστοιχο με την συμφωνία TTIP. Κύριε Ντεμαρτή, τι διδάγματα πραγματικά άντλησε από αυτό η Κομισιόν. Είναι ε, σαφές το ότι ναι πρέπει να δώσετε έμφαση στην ανάπτυξη, στις σε όλα τα καλά πράγματα. Ε, σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική σίγουρα μάθατε πολλά. Αλλά μάθατε τίποτα ουσιώδες υπό την έννοια ότι πρέπει πραγματικά και να των πολιτών εκπροσωπείται, να συμμετέχει, τα συμφέροντα των πολιτών εκπροσωπούνται. Ε, το ότι η άκτα δεν προχώρησε σας ε, ε, έκανε να αναγνωρίσετε ότι κάνατε κάποια λάθος προσέγγιση και πρέπει να αλλάξετε ίσως ε, προσέγγιση λοιπά. Δεύτερον, ένα αρνητικό, καθαρά αρνητικό στοιχείο. Είναι αυτή η επέκταση του ISDS ε, για τη ΣΥΤΑ, ε, τη συμφωνία αυτή τη γενική, θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το σχέδιο κειμένου ή τα σχέδια κειμένων που θα δίνουν τη δυνατότητα σε αμερικανικές επιχειρήσεις να μηνύουν κυβερνήσεις και αντίστροφο. Ακόμη και για την υλοποίηση αλλαγών στην νομοθεσία μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας ε, ΣΥΤΑ. Άρα πρόκειται για επίθεση όχι μόνο στα ε, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και στα πολιτικά. Θα μπορούν δηλαδή να επιβάλλουν επιχειρήσεις σε ό,τι θέλουν στις κυβερνήσεις ενδεχομένως. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση. Τώρα σε ό,τι αφορά το TTIP, τη συμφωνία TTIP, κάποια ε, σχόλια θα μπορούσαν να πούν ίσως και την άποψή τους ε, τα μέλη. Τι αντιπροσωπεύει η αναστολή των συνομιλίων για το τύπ. Την αντίληψη ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, δημόσια πίεση, πίεση από την κοινή γνώμη, πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις. Και πόσο πραγματική είναι αυτή η δέσμευση για δημόσιες διαβουλεύσεις. Είναι θέμα χρονοδιαγράμματος, Δηλαδή μήπως θέλουμε να αποφύγουμε να είναι ένα μείζον θέμα ε, της προεκλογικής εκστρατείας, να ξεπεράσουμε δηλαδή το εμπόδιο των ευρωεκλογών και να ξανασχοληθούμε μετά. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω τις απαντήσεις σας. Και τέλος, ένα δίδαγμα που αντλήσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια είναι η ανάγκη να γίνονται ανεξάρτητες, γνήσια ανεξάρτητες μελέτες αντικτύπου. Οι συζητήσει για το τίτλο, ο κύριος το επίτροπος, έρχεται εδώ και μας μιλάει για την ανάπτυξη, για τις τέσσερις εκατομμύρια θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια ευρώ ανάπτυξη. Και αυτά τα λένε και τα ξαναλένε και όλες οι εθνικές κυβερνήσεις. Και όταν σκάψει κανείς πιο κάτω, δεν υπάρχουν και τόσα πολλά. Ο συντάκτης ε, της έκθεσης ε, στη Γερμανία, της οποίας ε, ακούγονται και πολλά, λέει ότι ναι, δεν θα υπήρχε αρνητικός αντίκτυπος σε ό,τι αφορά την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θα, θα είναι πολύ λίγη η βελτίωση. Μήπως τελικά τα παραφουσκώνει η Κομισιόν τα πράγματα. Μήπως πρέπει να αντλήσετε και από εκεί ένα δίδαγμα. Να έχετε δηλαδή έναν ανεξάρτητο φορέα ε, που θα είναι σε εξέχουσα θέση και θα μπορεί να δίνει ε, ανεξάρτητες εκτιμήσεις ε, και αξιολογήσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Mm. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημαρτή, έχετε το λόγο. Yeah, thank, So, um, uh, Uh, uh, uh, Είμαι έτοιμος να προσπαθήσω να απαντήσω πολλέ ερωτήσει. πολλές ερωτήσεις. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επιλέξουμε διάφορα είδη ερωτήσεων που Το θέμα το... της επιβολής του νόμου και της σχέσης με το εμπόριο είναι σαφές καταρχήν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι σημαντικό τμήμα των εμπορικών συμφωνιών μας. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν μπορεί να είναι το μόνο εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μέσο, αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε από μια εμπορική συμφωνία να ε, πετύχει να μας φέρει τον ουρανό μετάστρα. Προσπαθούμε να περιλάβουμε το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης της εμπορική μας αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι περιορισμοί στις φιλοδοξίες και στο περιεχόμενο του κεφαλαίου, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι οι, ίδιε οι ίδιες οι αναπτυσσόμενες χώρες, διότι θέλουν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Για όλα αυτά είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Και θα ήθελα να επανέλθω για παράδειγμα ο κύριος Λάγκε πήρε το παράδειγμα των οικονομικών ε, συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Αυτό που λέμε ρήτρα εκτελεστική που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει αναστολή της συμφωνίας, η ανάκληση της συμφωνίας, αν υπάρξουν προβλήματα ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι μία από τις δυσκολίες που έχουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και εδώ Προσπαθούμε να βρούμε μια συμβιβαστική για όλα αυτά. Ας πούμε, σε αναφορά με την ε, Συμφωνία Κοτονού που αναφέρθηκε. Και αυτό έγινε και με την πρόσφατη συμφωνία με την ECOWAS ε, με την ε, Δυτική Αφρική. Και εδώ πάλι σίγουρα υπάρχει ένα θέμα σαφήνειας στόχου, ισορροπίας και σεβασμού για τον εταίρο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε. Για παράδειγμα, αναφέρθηκαν κάποια θέματα στον ΠΟΕ που αφορούν την ασφάλεια στα τρόφιμα, ε, ας πούμε για τους εκπροσώπους των ε, εκκλησιών ακούμε και πάλι ότι το εμπόριο δεν ήταν θετικό για την ανάπτυξη. Αντίθετα, τι είδαμε στον Παλί, επικράτησε ομοφωνία ανάμεσα στι αφρικανικές χώρες, τις ΑΚΕ και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να επιτύχουν καλή συμφωνία για την διευκόλυνση του εμπορίου, γιατί γνωρίζουν ότι η διευκόλυνση του εμπορίου είναι καλή για αυτούς. Και είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Και έρχονται σε σύγκρουση με την Ινδία σχεδόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν, υπά... δεν είναι θεμητός ο στόχος όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά αυτό το θέμα της ε, ασφάλειας στα τρόφιμα θα πρέπει να το διχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ε, δημιουργήσει, να μην προκαλέσει ανασφάλεια στα τρόφιμα αλλού. Και αυτό μόνο και μόνο το λέω για να σας πω ότι υπάρχει περιπλοκότητα όσον αφορά την επιβολή του συστήματος. και, την επιβολή των κυρώσεων, γιατί δεν χρησιμοποιούμε προσέγγιση κυρώσεων, ή δεν θεωρούμε πως αρκεί μια τέτοια προσέγγιση. Προτιμούμε να δουλέψουμε με συνεργασία και διάλογο με την κοινωνία των πολιτών από όλες τις πλευρές και πραγματικά όσοι εργάζονται με τα συστήματα των κυρώσεων, όπως είπα ας πούμε, στο κεφάλαιο το εργατικό δικαιωμάτων κτλ. Δεν λειτουργεί δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν οποιαδήποτε κύρωση οπουδήποτε, διότι ο τρόπος για την ενεργοποίηση των κυρώσεων ε, είναι, είναι πολύ δυσεφάρμοστος. Πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε σοβαρά υπόψη το θέμα των συμβάσεων ε, του ILO και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε όλα αυτά να ληφθούν υπόψη τις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις. Αλλά και πάλι λέω ότι δεν μπορούμε να ζητάμε να αντικαταστήσει ναι, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις όλες τις άλλες ε, ε, ε, ενωσιακές πολιτικές. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα ISDS που αναφέρθηκε από κάποιους. ISDS και ανησυχία για αυτό που ορισμένοι αποκαλούν επέκταση του ISDS ή το κινδύνους του ISDS της ΣΕΤΑ. Υπάρχουν πάνω από 500 διμερείς συμφωνίες ανάμεσα σε κράτη-μέλη και, και άλλα κράτη ε, όπου υπάρχει το ISDS και ποτέ δεν έχουμε ακούσει καμιά συζήτηση γι' αυτό. Αυτό που κάνουμε λοιπόν μετά την Λισαβόνα είναι η κοινοτικοποίηση αυτού του είδους του μέσου αλλά με ισορροπημένο τρόπο, με βελτίωση αυτού και δίνοντας τη δυνατότητα να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στην ρύθμιση, γιατί αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι είναι πολύ προσφυλές ε, να διατηρήσουμε το δικαίωμα ε, να, να ρυθμίζουμε εμείς και θα μιλήσω γαλλικά προς τον κύριο Ζαντό. Όχι, δεν διαπραγματευόμαστε επιλογές κοινωνικές. Δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε παζαρέματα με, με οποιονδήποτε εταίρο, ακόμα και αν είναι πολύ σημαντικός για να διαπραγματευτούμε τις δικές μας επιλογές τις κοινωνικές. Υπάρχουν ε, συλλογικές προτιμήσεις τις οποίες σεβόμαστε και αυτές θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και από τους εταίρους μας. Δεν θα διαπραγματευτούμε τις δικές μας βασικές ε, ρυθμίσεις, την προστασία του καταναλωτή, της υγείας μας, όχι. Δεν το πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Αναφέρατε, ε, μάλλον ρωτήσατε αν ε, η αδειοδότηση του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού 1507 είναι καλή ή κακό νέο για τις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Εγώ θα σας απαντήσω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σημαίνει απλά ότι εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία μας τελεία και παύλα. Η νομοθεσία αυτή υπάρχει, είναι εφαρμοστέα και εφαρμόσιμη και η απόφαση αυτή ελήφθη σε ιδιαίτερες περιστάσεις και αυτό που διακυβεύεται στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ δεν είναι η αμφισβήτηση της δικής μας νομοθεσίας για τους γεννητικά τροποποιημένους οργανισμούς που θα εξακολουθήσει να ισχύει ως έχει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε θέματα καλλιέργειας των γάμματα φόμικρων υπάρχει μεγάλη αντίρρηση από πλευρά τη κοινή γνώμη στην Ευρώπη και θα συνεχιστεί και δεν θα διαπραγματευτούμε με τη ΣΥΠΑ τη δυνατότητα να επεκταθούν οι δικέ μα καλλιέργειε εφόσον οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν το επιθυμούν. Δεν είναι αυτό στοιχείο τη διαπραγμάτευση. Δεν πρόκειται δηλαδή να εισάγουμε ούτε κρέα με ορμόνε. Ακούω να γίνεται λόγο γι' αυτό. Όχι, καθόλου. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τι επιλογέ μα, να αναπτύξουμε όμως μια προσέγγιση με τους μεγάλους μας εταίρους και με τις είπα, δηλαδή που θα επιτρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία και η απασχόληση προσπαθώντας να έχουμε και καλύτερη σύγκληση ρυθμιστική αλλά χωρίς να αμφισβητήσουμε και άλλη μια φορά τις δικές μας επιλογές. To, ε, ε, ε, English, on, public services. Θα επανέλθω στα αγγλικά για τις δημόσιες υπηρεσίες. Και εδώ θα είμαι σαφής. Δεν διαπραγματευόμαστε με οποιοδήποτε τρίτη χώρα, εταίρο, για τις δημόσιες μας υπηρεσίες. Υπάρχει σαφής πρόβλεψη στην ΓΑΤ για τις δημόσιες υπηρεσίες Όποια και να είναι η επιλογή στις διαπραγματεύσεις, είτε αρνητικός κατάλογος είτε θετικός κατάλογος, που μετά μπορεί να μετατραπεί σε αρνητικό, πάντως αυτές οι διατάξεις GATT, αυτή η διάταξη μάλλον, έχει επανεισαχθεί ως είχε στο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες και στο παράρτημα 2 αυτού του κεφαλαίου που σημαίνει ότι αυτές οι διατάξεις υπάρχουν και με συγκεκριμένο χώρο για την πολιτική και το ίδιο για το νερό. Ε, και πολλά πράγματα ακούγονται δεξιά-αριστερά στο δημόσιο χώρο, αλλά αυτά όλα δεν αντιστοιχούν σε αυτό που εμείς κάνουμε. Και με τη ΣΥΠΑ το ίδιο ισχύει. Βεβαίως δεν λέω ότι οι ΕΠΑ θα χαρούν όλα αυτά, Πάντως δεν τίθεται θέμα διαπραγμάτευσης. Και πάλι λοιπόν θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα ως έχει και να διαπραγματευτούμε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες με βάση τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και όχι σαν κάτι που είναι ένα ιδεολογικό πρόγραμμα, όραμα, δεξιό, αριστερό κτλ. Όχι. Είναι κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις απασχόληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ πασίγνωστο και τεκμηριωμένο ότι οι θέσει απασχόληση που συνδέονται με το εμπόριο είναι καλύτερα αμοιβόμενε από άλλε θέσει. Αυτό είναι σαφέ. Δεν είναι δύσκολο να το δει κανεί και στι αναπτυσσόμενε χώρε ότι οι χώρε που είναι ανοιχτέ στο εμπόριο λειτουργούν καλύτερα, αποδίδουν καλύτερα όσον αφορά την μείωση τη φτώχεια. Ε, όλα αυτά είναι ορατά. Και αυτή είναι η ε, κατεύθυνση που ακολουθούμε. Και τα τελευταία σχόλια... Τελευταία ε, ερώτηση εξαγωγικές ε, αποζημιώσεις στην, για τη Γεωργία δεν υπάρχουν πλέον μετά από την τελευταία μεταρρύθμιση θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιπτώσεις κρίσης και ειλικρινά πιστεύω πως δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε σε περιπτώσεις κρίσης γιατί σημαίνει ότι θα εξάγουμε την κρίση μας αλλού. Οπότε δεν νομίζω πως είναι πολύ πιθανό να ξαναχρησιμοποιηθούν οι επιστροφές στις εξαγωγές. Και έγινε και μια ανακοίνωση για την Αφρική ε, για όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τι κάνει η Ένωση, αλλά και τι κάνουν και οι άλλοι. Διότι δεν είναι μόνο θέμα εξαγωγών, ανταγωνισμού στην... Ε, δεν είναι μόνο θέμα των επιδοτήσεων στις εξωγές, είναι και το θέμα της επιδότησης των, πιστώσεων, των εξαγωγικών πιστώσεων, από ορισμένους, ας πούμε, τους είπα, ή τη χρήση του, ε, της, της, της, της βοήθειας σε είδος Πώ δηλαδή οι κρατικέ επιχειρήσει χρησιμοποιούνται με άδικο τρόπο, για παράδειγμα από την Κίνα, και επηρεάζουν τι αγορέ. Και βεβαίω αν τα δει όλα αυτά κανεί σε ένα παγκόσμιο πακέτο, βλέπουμε ότι και άλλοι κάνουν προσπάθειε και άλλοι και είμαι βέβαιο ότι σε κάποια φάση θα είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε και να να μην το ξανακάνουμε. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, διότι ούτε και οι άλλοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν αντίστοιχε δεσμεύσει. Και πάλι λοιπόν ας δούμε ε, τις ευρύτερες προοπτικές για την ναύτα. Για την άκτα, συγγνώμη, άκτα. Ε, ο κ. Μέρφυ έφυγε, αλλά κάποιο θα του πει την απάντησή μου, φαντάζομαι. Θα το αναφέρει την απάντησή μου. Η απάντησή μου λοιπόν είναι η εξή. Πρώτον, Υπάρχουν διάφορα δάγματα που καρίσει κανείς να αποκοπήσει από την άκτα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει να συμμετέχουμε, όχι γιατί ήταν διά, του διαόλου, αλλά γιατί τη προστιθέμενη αξία αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν πολύ περιορισμένη. Και τελικά δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσε για μας και είναι μια διαπραγμάτευση όπου δεν αναλάβαμε δεσμεύσει. είναι μια διαπραγμάτευση που ξεπερνούσε τη δική μας κοινωτική νομοθεσία, δημιούργησε πολλές συγκινήσεις, υπάρχουν διδάγματα για, όσον αφορά την διαφάνεια και τα έχουμε χρησιμοποιήσει για τις διαπραγματεύσεις για τη TTIP και θα περάσουμε από την άκτα στη διαφάνεια. Να θυμίσω ότι για τη διαφάνεια κάνουμε πάρα πολλά στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Θα σας πω ότι προέρχομαι από τον Εθνικό Διοικητικό Μηχανισμό. Εργάζομαι στην Κομισιόν εδώ και 25 χρόνια. Και αν συγκρίνω ποια είναι η διαφάνεια ενός εθνικού διοικητικού οργανισμού και της Κομισιόν, πραγματικά δεν έχουμε να ντραπούμε για τίποτα. Να είμαι πιο συγκεκριμένο στο τι κάνουμε για την TTIP. Πρώτον, δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά ένα σύνολο αρχικών ε, ε, ε, γράφων που περιλαμβάνουν τις θέσεις μας και το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Έχουμε μια ανεξάρτητη μελέτη για να αξιολογήσουμε τον δυνητικό αντίκτυπο και να πω ακριβώς τι κάνουμε με την αξιολόγηση αντίκτυπου. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να περιλαμβάνει περισσότερες αξιολογήσεις αντικτύπου από ότι η DG Trade. Έχουμε τεσσάρων αξιολογήσεις, μάλλον συγγνώμη, τέσσερα βήματα στην αξιολόγηση. Έχουμε την SIS, δηλαδή ε, η, αξιολόγηση βιώσιμου αντίκτυπου, έχουμε ε, την πρώτη αξιολόγηση και έχουμε και εξπόστα αξιολόγηση που γίνεται για κάθε μια πολιτική. Αλλά τα δύο στοιχεία, τα μεσαία, δεν χρησιμοποιούνται σε καμιά άλλη πολιτική. Δεν υπάρχει SIA για καμιά άλλη πολιτική, ούτε οικονομική ανάλυση στην ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη συμφωνία ή μια συγκεκριμένη νομοθεσία ανάμεσα στους δύο, τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής. Δεν έχουμε τίποτα να ντραπούμε λοιπόν ε, και χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα ε, πρότυπα ε, για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των των μέτρων μας. Ε, δεν ε, πρόκειται για, για ε, καμιά μπανανία δηλαδή, ούτε για παραμύθια. Πρόκειται για πραγματικές ε, μελέτες, εξολογήσεις και είναι σαφές ότι είμαστε πολύ εντάξει. Επίσης κάνουμε και πριν και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δημόσιες διαβουλεύσεις Έχουμε πολλούς ε, εμπειρογνώμονες και περιβαλλοντικούς ε, που συμμετέχουν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 160 εμπλεκόμενοι φορείς ήταν ε, παρόντες σε μια δημόσια δίπλωση που είχαμε. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε. Αλλά βέβαια στόχος μας είναι και να ενημερώνουμε τα κρατημέλη και το κοινοβούλιο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, διότι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία και των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών. Ε, είμαστε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μας ελέγχουν. Έχουμε το νομοθετικό σώμα, το κοινοβούλιο και το συμβούλιο που μας ελέγχουν. Αυτό γίνεται σε κάθε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και βέβαια, να υπενθυμίσω ότι ο Ευρωπαϊκό ε, Διαμεσολαβητή τον Ιανουάριο είπε ότι είμαστε πιο ανοιχτοί σε σχέση με το παρελθόν για αυτά τα θέματα και οποιαδήποτε συμφωνία ε, θα είναι δυνατόν να ελεγχθεί σε όλες τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσουμε στην έγκριση. Οποιαδήποτε συμφωνία λοιπόν θα είναι αφόσον ε, υπογραφεί στη διάθεση των πολιτών. Δεν είμαι βέβαιος βέβαια ότι θα μπορέσουν όλοι οι πολίτες ε, ε, σίγουρα να κατανοήσουν το περιεχόμενο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξηγήσουμε στους πολίτες τι συμβαίνει. Και σας υπερθυμίσω τη σχετική μας δέσμευση. να απαντήσω πάλι στα γαλλικά, στα ερώτημα του κυρίου Ζαντό. Εσωτερική συνεκτικότητα και συνέπεια των εμπορικών μας διαπραγματεύσεων. Υπάρχει σχέση μεταξύ των διαφόρων εμπορικών διαπραγματεύσεων και των εμπορικών διαπραγματεύσεων και των άλλων πολιτικών. Φυσικά, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε και να αποκομίσουμε όφελο από αυτέ τι εμπορικέ διαπραγματεύσει ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία και την ανάπτυξη, υπάρχουν ορισμένε προποθέσει. Πόσο ανταγωνιστικοί μπορεί να είμαστε, πόσο παραγωγικοί μπορεί να είμαστε. Και βέβαια, συμφωνώ, δεν είναι μόνο θέμα εξαγωγών, αλλά και εισαγωγών. Το global value chain, δηλαδή η συνολική αλυσίδα αξίας δεν είναι αμεληταίο ε, το κομμάτι των εισαγωγών. Πρέπει να ε, βλέπουμε τα πράγματα συνολικά και όχι μερκαντιλιστικά. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε ξεχωριστά τις εξαγωγές από τις εισαγωγές. Φυσικά και μπορούμε να βελτιωθούμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας ε, την συνέπεια. Να, και να είμαστε συνέπειες, δεν ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Εξωτερική συνέπεια συνεκτικότητα. Μιλήστε για τον κύριο Ντεφρέιν. Δεν ήταν ποτέ ούτε προκατοχό μου ούτε στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ήταν γενικό διευθυντή στη διεύθυνση των εξωτερικών σχέσεων και επικεφαλή του γραφείου του κυρίου Λαμή σε ένα κομμάτι τη θητεία του. Φυσικά και έχει δικαίωμα να λέει τι απόψει του ο κύριο Ντεφρέιν, όπω και οποιοδήποτε άλλο βέβαια. Είναι σαφές ότι δεν ε, είμαστε στο ίδιο μήκο ε, δεν έχουμε τι ίδιες η συμφωνία TTIP παρέχει ευκαιρίες. Για μας δεν είναι ιδεολογική προσέγγιση, ούτε υπέρ ούτε κατά της Κίνας. Δεν είναι πολιτική συγκράτηση ε, παρεμπόδισης της Κίνας. Για κάποιους μπορεί, αλλά δεν είναι δική μας πολιτική. Και έχουμε και για τις επενδύσεις διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε πιο πολλά πράγματα κάποια στιγμή με την Κίνα. Αλλά δεν είμαστε αφελείς ούτε με την Κίνα ούτε με τη ΣΥΠΑ. ούτε εκφράζουν κάποια ιδεολογική προτίμηση υπό την μία την άλλη έννοια. Είναι σαφές ότι για μας η αμερικανική οικονομία είναι σίγουρα πιο ανοιχτή από την κινέζικη. Αυτά είχα να πω. Λυπούμε που μακρηγόρησα και δεν τα είπα έτσι και με τη σειρά. Ίσως ξέχασα, σίγουρα ξέχασα μερικά, αλλά σας ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά γι' αυτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε να κάνω τρεις προσωπικές παρατηρήσεις. Πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Και νομίζω ότι υπάρχουν διόψεις της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Επιτροπής μας με την Κομισιόν. Πρώτον, δύο οργανικές σχέσεις. Υποδειγματικές ήταν εν γέννη αυτές οι σχέσεις Είχαμε πολύ υψηλά επίπεδα ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωση. Ήμουν εισηγητή για τη συμφωνία TTIP και εύχομαι στο Καπιτόλιο ο ομόλογο μου να είχε την ίδια πρόσβαση που είχα εγώ στι πληροφορίε. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αλλά ισχύει και για τα άλλα μέλη τη Επιτροπής Παρακολούθησης ε, της Επιτροπής μας στο TTIP. Φυσικά και είμαστε υπεύθυνοι και για το επιτεύγμα αυτό. Θα πρέπει όμως να συγχαρούμε και την Κομισιόν, να την επενέσουμε, διότι πάντοτε ήταν έτοιμη να έλθει εδώ να απαντήσει στα αιτήματα, στις απαιτήσεις μας, τα έλεγα ακόμη και στις διαταγές μας εντό αγωγικών. Και να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να γραφεί στα πρακτικά. Η Κομισιόν δεν θέτησε ποτέ τη καμία δέσμευση απέναντι στη δική μα επιτροπή. Οτιδήποτε δεσμεύτηκε να κάνει το έπραξε. Τουλάχιστον προσπάθησε να το πράξει. Και με πολύ θετικό τρόπο και με πολύ επέφθενο τρόπο. Δεύτερη παρατήρηση πολιτικού χαρακτήρα. Πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας, η εμπορική πολιτική αποφασιζόταν από Κομισιόν και Συμβούλια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα ουσιαστικό. Γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, ε, συζητήσεις. Αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονταν από τα άλλα δύο όργανα. Με τη συνδίκη της Λισαβόνας άλλαξαν τα πάντα. Και έτσι πήρε σάρκα και όχι μονοστά ε, η συνθήκη της Λισαβόνας. Και πράγματι πετύχαμε και γιατί μπορούσαμε και γιατί αγωνιστήκαμε γι' αυτό αλλά και γιατί δεν αντιστάθηκε η Κομισιόν. αντιθέτω, ήταν έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί μας. Ήδη και από τότε που σχεδόν ήταν η μόνη αρμόδιοι για αυτό το τομέα. Σε αυτή την πενταετία, λοιπόν, με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τι πρωτοβουλίες της Κομισιόν με μια-δυο εξαιρέσεις. Αναφέρθηκε η μία, ήταν η άκτα. Ήταν ένα από τα μείζωνα συμβάντα ε, της πενταετίας αυτής. Με την ίδια την πλειοψηφία με την οποία απορρίφθηκε η άκτα, εγκρίθηκαν όλες οι άλλες συμφωνίες από αυτό το ίδιο κοινοβούλιο και από αυτήν την Επιτροπή. Τέλος, ένα θέμα ουσίας που αφορά και την κατεύθυνση της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Τα εμπορικά ανοίγματα δεν είναι διακριτική νεοφιλελεύθερη απόφαση που λαμβάνει η Κομισιόν. Είναι συνταγματική εντολή. Το λένε οι συνθήκες. Το λέει το άρθρο 3 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 206 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το λέει free and fair trade, ελεύθερο και δίκαιο ε, εμπόριο. Δεν είναι δογματικές εκφράσεις, είναι συνταγματική αρχή. Το άνοιγμα του εμπορίου, κατάργηση, κατάρριψη των εμπορικών φραγμών είναι ε, θεσμική, είναι συνταγματική εντολή που δίνεται από τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και το άρθρο 21 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να σεβόμαστε και να τηρούμε την εντολή μας από το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 206 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που με κάνει ιδιαίτερη περήφανο ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια εμπορική πολιτική της Ένωσης που να είναι αξιόπιστη, προβλέψιμη, αποτελεσματική και την εκπροσωπούν ε, και την ε, προσυπογράφουν ε, πολιτικές ομάδες. Υπήρξαν κάποιες βέβαια που δεν θέλησαν να την υποστηρίξουν. δεν θέλησαν να στηρίξουν τις κρατούσες απόψεις εδώ ούτε στο κοινοβουλίο στην Ένωση. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Ίσως είμαι από μέσα τις πολιτικές ομάδες που δεν ε, μας στηρίζουν, αλλά όταν θα διαπραγματευτούμε με τρίτες χώρες έχουμε αυτό το πλονέκτημα γιατί ξέρουν αυτές οι χώρες ότι Μπορεί τα κοινοβούλια να έρχονται και να φεύγουν και η Κομισιόν μπορεί να έρθει και να φύγει και το Συμβούλιο μπορεί να αλλάξει, αλλά η εμπορική πολιτική της Ένωσης θα παραμείνει. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι. Ευχαριστώ πολύ. Uh, this uh, the uh, Τώρα προχωρούμε στο τμήμα της συνεδριάσεως που θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών και θα παρακαλέσω εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που έχουν το δικαίωμα ή και το καθήκον να παραμείνουν, οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν.